Καλησπέρα σα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι έχει άδειε θέσει. Μπορούν να καθίσουν οι καλεσμένοι Μα Δεν είναι ανάγκη να στέκονται όρθιοι. Θέσεις υπάρχουν. Παρακαλώ, καθίστε. Ακυρίσω την έναρξη της Επιτροπής Γεωργίας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξή μας. Ο κύριος Άγνη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Δεν ακούμε διερμηνή από τα αγγλικά, κύριε Πρόεδρε, ούτε εγώ ούτε άλλος συνάδελφος που παρακολουθεί την αγγλική καμπίνα, την αγγλική διερμηνία. Μήπως ξέχασα να πατήσουν το μικρόφωνο οι στην αγγλική καμπίνα. Για, αλέξτε το παρακαλώ. Okay. Moment, we should give time for. It's okay. Εντάξει τώρα. Ωραία. Έχουμε αναμετάδοση από το διαδίκτυο της σημερινής συνεδρίασης. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά την σημερινή μας συνεδρίαση, μετά το πέρας της συνεδρίασης μας από απογευματινής, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε τα αγγλικά. Όπως είπα, έχουμε αναμετάδοση από το διαδίκτυο της συνεδρίασής μας. Ah, Και με τα γερμανικά υπάρχει πρόβλημα, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να διορθωθεί το τεχνικό πρόβλημα. Chairman, yes, the problem we seem to be getting is that we get a bit of English. Ακούμε λίγα αγγλικά, μετά ακούμε λίγα γερμανικά μπερδεμένα. Μάλλον υπάρχει ένα πρόβλημα στα κανάλια. Τι μας παίζει κανείς για προχριστουγεννιάτικα παιχνίδια. Όχι, ας δώσουμε την ευκαιρία στον τεχνικό μας να διορθώσει το πρόβλημα. Διορθώθηκε το πρόβλημα. We όχι, πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Okay. Για τρία λεπτάκια διάλειμμα. Thank <laughs> you. Ο κύριος Άγνιο μας διαβεβαιώνει ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν διερμηνή αγγλικά, γερμανικά, χωριστά. Κύριε Νόεχλ, ακούτε τη γερμανική διερμηνία. Ωραία. Έχουμε και γερμανική διερμηνία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ή μάλλον να συνεχίσουμε. Είπαμε ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση και να σας υπενθυμίσω ότι στις 6.30 μετά το πέρας της συνεδρίασης θα έχουμε μία σεπτή χριστουγεννιάτικη δεξίωση και ε, να περάσουμε στην ενημέρωση που μας κάνει η κυρία Νταντσίλα για τα αποτελέσματα του τριμέρους διαλόγου. Ήθεστε να ενημερώνετε η Επιτροπή από τον αρμόδιο εισηγητή. Ο κύριος Αντρια είναι ο συντονιστής μας. Οπότε θα ήθελα είτε ο συντονιστή είτε η κυρία Νταντσίλα να μας ενημερώσουν για, το, για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου και να μας κάνουν και τις προτάσεις τους. Ο κύριος Ανδρία, Ευχαριστώ. Δυστυχώ η κυρία Νταντσίλα κολλείεται, είχε ανηλυμένε υποχρεώσει στη Ρουμανία και μου ανέθεσε να σα ενημερώσω εγώ για τα αποτελέσματα του πρώτου ημερού διαλόγου για τις ενοποιημένες στατιστικές πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μάλιστα έχει οριστεί και ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα από τους ε, εκπροσώπους μας στη διαπραγμάτευση και θέλουν μόνο σε δύο τριμερείς διαλόγους να διεκπεράσουν το θέμα και να καταλήξουν συμφωνία. Και μάλιστα στον πρώτο τριμερή διάλογο της περασμένης εβδομάδας ήδη είχαμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ιδού ε, η επιτυχία, το επιτυχημένο αποτέλεσμα που επέτρεψε συμφωνία σε αρκετά σημεία που θα σας παρουσιάσω. Άρα θα υλοποιήσουμε το στόχο μας. Άρθρο 2 για τους ορισμούς, ιδιαίτερα για την ε, ωφέλιμη γεωργική ε, επιφάνεια. Επίσης άρθρο 3 για το πεδίο εφαρμογή ε, της τροπολογίας υπερθμών 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διευκρίνει το στόχο μεταξύ το το στόχο κάλυψε 88% και τα ελάχιστα κατόφλια του άρθρου 6. Ε, Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 για τις πηγές των δεδομένων και το 5α για τη χρήση των μητρών των φορέων πληρωμής ε, έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ε, διαφόρων εισηγητών. Και μια και το άρθρο 4 εξασφαλίζει πρόσβαση στις πληροφορίες, το 5α που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσύρθηκε γιατί κρίθη πλέον περιττό. Α, τροπολογία 22, δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποσυρθεί. Τέταρτο σημείο. Μετά τις διευκρινήσεις για το άρθρο 11, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δειγμάτων και των στοιχείων, των δεδομένων, οι εισηγητέ έκριναν ότι, το άρθρο, ότι η τροπολογία 23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύπτεται από τα μέτρα τα προληπτικά. Σε ό,τι αφορά την αρχή της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης, τη υποχρεωτική και αυτό έγινε δεκτό, δηλαδή η τροπολογία 33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και η τροπολογία 16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν δεκτέ. Εξασφαλίζουν τη σύνδεση αυτού του κανονισμού με το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης ένας εκτενής κατάλογος τεχνικών διορθώσεων εγκρίθηκε καθώ και τα δύο παραρτήματα, τα υπαριθμών 4 και 5 μετά τον πρώτο τριμερή διάλογο ε, είχαμε συζήτηση και για τα πιο αγαθόδη σημεία, δηλαδή το άρθρο 8 των τεχνικών διευκρινήσεων για τους διάφορους τρόπους και το άρθρο 9 για τα ad hoc modules. Και τα τρία μέρη παρουσίασαν τις προτιμήσεις τους και η τεχνική ομάδα θα επιληφθεί του ζητήματος προκειμένου να προτείνει κάποιες λύσεις ε, στον επόμενο τριμερή διάλογο και άλλα θέματα παραπέμφθηκαν στην τεχνική ομάδα για να αναδιατυπωθούν εν ώψη τη τελική συμφωνία. Και στον επόμενο τριμερή διάλογο, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο τελευταίο, θα γίνει στο Στρασβούργο 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Και μάλιστα θα προηγηθεί η συνεδρία των σχεδόν εισηγητών από τι 2 το απόγευμα. Και πάλι η εισηγήτριά μα, η κυρία Ταντσίλα, που ζητά συγγνώμη για την απουσία τη. Ε, σα διαβεβαιώνει ότι η βοηθή τη. Ε, που είναι παρόντες είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε απορίες σας και να διασκεδάσουν τις ανησυχίες σας. Αυτά επί των ολοκληρωμένων στατιστικών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ε, μια έκθεση της κυρίας ε, Βιόριτσα Νταντσίλα. Μάλιστα, περνάμε στη συζήτηση. Το λόγο έχει πρώτος ο κύριος Άγνιου. Thank you, ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή αφορά στατιστικές γεωργικές και αναφέρει μια έρευνα δομημένη που αποβλέπει να συλλέξει τα δεδομένα. Την περασμένη πέμπτη έλειπα στη συνάντηση με την Επιτροπή, αλλά θέλουμε τώρα να αποκεντρώσουμε το όλο σύστημα και αυτό πώς θα το συνδέσουμε με αυτό που είπαν. Ευχαριστώ. Κύριος Λουαζό. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία εισηγήτρια αποσιάζει. Νομίζω δεν έχουμε κάνει στατιστικέ και τον τρόπο συλλογή σε σχέση δηλαδή, με τη βελτίωση της, των συνδικών για του γεωργού. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι στο μελλοντικό γεωργικό σύστημα θα, στατιστικό θα πρέπει να αυξήσουμε τι ε, προτεραιότητε. Τώρα θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο. Κάποιες χώρες είδαμε πρόσφατα, όπως η Γαλλία, αντιμετώπισαν απώλειες ε, θέσεων εργασίας και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική, διορατική για την κλιματική αλλαγή. Να αντιμετωπίσουμε την εξαιρεσία και να δώσουμε αποζημιώσεις όπου θα χρειαστεί, αρκετά δηλαδή. Πρέπει να μιλήσουμε επίσης και για μια δίκαιη αγορά Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα για να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και τον αθέμητο ανταγωνισμό και πώς θα το κάνουμε αυτό, αναρωτιέμαι. Θέλετε να είμαστε πιο ισχυροί στην διεθνή σκηνή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις αγορές, τις εξαγωγές, χωρίς να μειώσουμε ε, τους ε, φραγμούς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε επίσης τι γίνεται και με τα θέματα διατροφής. Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένου τομεί ώστε να έχουμε ε, αυτάρκεια διατροφική. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να είναι τα κύρια σημεία που θα πρέπει να εξετάσουμε στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νόιχλ. Äh, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και εγώ της Μαρία Χόιμπουργκ. Η κυρία Χόιμπουργκ και εγώ ασχοληθήκαμε με την ε, έκθεση όσον αφορά τη στατιστική και οι δύο παρατηρήσαμε ότι επιγόντως χρειαζόμαστε ε, καταλόγους για τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ε, θίγονται και κυρίως να δούμε ε, σε, ποια, σε ποιες ομάδες εργαζομένων ανήκουν αυτές οι κατηγορίες. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ποιες επιχειρήσεις, ποιες εκμεταλλεύσεις ε, συμπεριλαμβάνονται. Το ελάχιστο μέγεθος πρέπει να οριστεί στα 4 εκτάρια σύμφωνα με την Επιτροπή. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αλλά να μην ε, παραβλέψουμε και τις μικρές. Κάτι θα ήταν λάθο. Τι χρειαζόμαστε και τι μικρέ γεωργικέ εκμεταλλεύσει, οι οποίε δεν πρέπει να είναι αόρατε ε, στην στατιστική. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, να, να ορίσουμε την δομή του holding και των εκμεταλλεύσεων και για τις μεγάλες και για τις μικρές εκμεταλλεύσει, χωρίς ελάχιστα και ανώτατα όρια. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Κυρία Σένρα, κυρία παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σύντομα, να τονίσω την ανάγκη προάσπισης της θέσης του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον ρόλο των γυναικών γεωργών στα πλαίσια των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Η θέση δηλαδή του Κοινοβουλίου όπως έχει αρχικά να διατηρηθεί και στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Είχαμε με αντάλλαγη απόψε να έχουμε κάνει δεκτή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγάλη πλειοψηφία, οπότε η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες επιβαρύνσεις για τους Γιώργους, που είναι όμως απαραίτητες για μια σωστή διαχείριση και των πληροφοριών. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμη η ενημέρωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντρία. Παρακαλώ διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας στην συγκεκριά μας, την κυρία Ταντσίλα. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 4, εκτός και αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Όχι, οπότε περνάμε στο σημείο 4 που θα ακούσουμε την παρουσίαση από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενός, της παρουσίας ενός σχεδίου ε, εφαρμοστικής ε, πράξης για τους κανόνες εφαρμογής της διαχείρισης του συστήματος δεσμολογικών προσωστώσεων χωρίς άδειες. Α, ο κύριος Αντρέ ζήτησε το λόγο για να κάνει κάποια σχόλια. Δύο λόγια για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη συζήτηση. Όντως, θα δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις τις οποίες σημείωσα, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στη θέση της ε, και όπως είπε ο κύριος Λαζό, οι στατιστικές ε, στόχο έχουν την ε, δημιουργία ενός στιγμιότυπου της πραγματικότητας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αφησιμία για το ρόλο των στατιστικών. Δεν επηρεάζουν ή προσανατολίζουν οι στατιστικές, απλώς μας δίνουν μια εικόνα της πραγματικότητας, ώστε στη συνέχεια έχοντας επίγνωση πραγματικότητας να προτείνουμε κάποιους πολιτικούς προσανατολισμούς. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία της κυρίας Νόιχλ που μας είπε ότι θέλουμε κάποια εργαλεία και σωστά μέσα για την ανάλυση των διαπιστώσεων και της διάγνωσης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έθεσαν ερωτήσεις. Θα σταλούν γραπτός οι απαντήσεις από την κυρία Νταντσίλα που είναι και η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα ε, της εκτελεστικής πράξης που, που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της διαχείρισης του συστήματος δεσμολογικών ποσοστώσεων ε, χωρίς ε, άδεια. Η κυρία Σραέρ Πύρικ, ε, η συντονίστριά μας, ε, ζήτησε την ενημέρωση αυτή. υπάρχει ένα επίπεδο, μια μείωση των δασμών που επιτρέπεται σε περιορισμένες ποσότητες εισαγωγών και αυτό λαμβάνει τη μορφή δεσμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγέ ιδιαίτερη ε, προέλευση στα πλαίσια του σύστηματος προνομιακών ποσοστώσεων. Ε, η διαχείριση του συστήματος δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται ε, κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή δηλαδή Επιτροπή. Εν βέβαια σε, ε, συναρμόδια είναι και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα θέματα αυτά. Για τις λεπτομέρειες θα μας ενημερώσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο και καλωσορίζω και του δίνω το λόγο για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Μπρούνο Βαρδάιερ. Παρακαλώ. Ε, thanks a lot, Chairman. Ε, yes. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε. Όταν η Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, όταν έχουμε ευαίσθητος τομείς παραγωγής, τότε δεν είναι και τόσο διατεθειμένοι η Ένωση να ανοίξει πλήρως την αγορά και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ποσοστώσεις, δασμολογικές ποσοστώσεις. Το οποίο σημαίνει ότι προτείνουμε μια περιορισμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά τον όγκο και με κάποιο έτσι, κάποια εφαρμογή έτσι, μιας λογικής ποσόστοσης. Συνήθως αυτές οι ποσοστώσεις είναι ατελείς, αλλά όχι πάντα. Έχουμε λοιπόν πάνω από 500.000 ποσοστώσεις οι οποίες εφαρμόζονται και που διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση από τις χώρες και την Κομισιόν. Πράγματι, έχουμε 350 ποσοστώσεις οι οποίες διαχειρίζονται από την ταξούτ με σειρά προσέλευσης όπως τη λέμε. και έχουμε άλλες 150 ποσοστώσεις που διαχειρίζεται η Γενική Διευθυνσία στα πλαίσια μιας ε, ταυτόχρονης εξέτασης, όπως τη λέμε. Έχουμε λοιπόν στα πλαίσια τη γενική μα διεύθυνση και μετά από την συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε μια, ένα διχωρισμό μεταξύ κατεξοδότηση και πιστική πράξη. Και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους ενδιαφερόμενους και τις χώρες μέλη, ώστε για αυτές τις 150 ποσοστώσεις να ακολουθούμε μία κατοξιζώση και μία εκκληστική πράξη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι σημαντικό να έχουμε δικασίες εναρμόνισης και απλούστευσης και αυτό που κάνουμε θέλουμε να το πετύχουμε σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δουλειά μας πριν περίπου τρία χρόνια μέσω ενό σεμιναρίου όχι από τις υπηρεσίες της Κομισιόν αλλά ενό σεμιναρίου με τις χώρες μέλη και με τους ενδιαφερόμενους όπου προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας και να χαράξουμε μια κοινή γραμμή αντιμετώπιση. Και οι χώρες μέλη, όπως και οι ενδιαφερόμενοι, είχαν σαφή προσέγγιση όσον αφορά την γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δηλαδή τόνιζαν το ότι το νέο κείμενο, η νέα Εκθεστική και νέα κατεξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να επικεντρώνεται στους ε, φορείς, τους οικονομικούς και θα έπρεπε ως τελικό αποτέλεσμα να έχουμε την αύξηση της διαφάνειας και τέλος το σύστημα που θα έχουμε στη διάθεσή μας προς εφαρμογή και διαχείριση να μην ε, προαγάγει την κερδοσκοπία Οπότε είναι εύκολο σχετικά αυτό κατά κάποιο τρόπο γιατί αυτές οι ποσοστώσεις ε, δεν είναι αντικείμενο μεγάλης ζήτησης και ε, δεν ζητούνται σε κάποιες περιπτώσεις κιόλα. αλλά σε κάποιες άλλες καταστάσεις η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε αυτό που ονομάζουν οι οικονομολόγοι μίσθωση ποσοστώσεων που είναι πολύ υψηλή. Δηλαδή έχουμε ένα όφελος για τον ενδιαφερόμενο ο οποίο έχει μια άδεια εισαγωγή σε σχέση με αυτή την ποσόστοση ένα τμήμα τη, και ε, βλέπουμε εκεί ότι το όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ υψηλό. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε αυτές τι περιπτώσεις και επειδή η ζήτηση είναι πολύ υψηλότερη από την προσφορά στα πλαίσια του ποσοστώσεων πάντα, τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε συντελεστή κατανομή. Εύκολο να το κατανοήσει κανεί αυτό έτσι. Α πούμε ότι έχουμε μια ποσόστοση χίλια και εμεί έχουμε μια ζήτηση για 2.000. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, τι κάνουμε, ο συντελεστή κατανομή θα είναι 0,5. Απλά μαθηματικά Όμω, σε άλλε περιπτώσει, ο συντελεστής κατανομή είναι πολύ χαμηλότερο. Ακόμα και πιο χαμηλό από το 1%. Οπότε Κυρίω για το σκόρδο σημαίνει, συμβαίνει αυτό σήμερα. Και το αντιμετωπίζουμε αυτό κάνοντας μια διάκριση μεταξύ του να αφιχθέντος αγωγία και του, του παλιού Οπότε έχουμε ένα 70% της ποσόστοσης, το οποίο πηγαίνει ας πούμε στους παραδοσιακούς εισαγωγή και ένα 30% που υπολείπεται πάει στον νεοαφιχθέντα, στον καινούριο εισαγωγέα. Και μετά από κάποια χρόνια και ο καινούριο γίνεται παλιός. Οι χώρες μένουν λοιπόν και ενδιαφερόμενοι δεν ικανοποιούνται πλήρω από αυτό το σύστημα όμως, το οποίο φαίνεται να δημιουργεί κάποιες αλλοιώσεις και να προκαλεί και κάποια ασφάλματα όσον αφορά την εφαρμογή του στις χώρες μέλη. Οπότε ζήτησαν λοιπόν οι χώρες μέλη μία τροποποίηση αυτού του συστήματος και αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς να κάνουμε. Όμως, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις η διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων ήδη είναι ενσωματωμένη στις πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις τρίτες χώρες. Και αυτό αφορά κυρίως τις περιπτώσεις ποσόστοσης για το κινέζικο σκόρδο και το αργεντίνικο σκόρδο. Σύμφωνα λοιπόν με τις ιδιαιτερότητες ή τις προβλέψεις αυτών των ημερών ή πολυμερών ε, συμφωνιών, τότε θα πρέπει είτε να κάνουμε συζητήσεις με αυτό το τρίτο μέρος, είτε ενδεχομένως να διαπραγματευτούμε νέα συμφωνία με αυτή την ε, τρίτη χώρα. Τώρα, όπου χρειάζεται και οι συνάδελφοί μας οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα διεθνή θέματα ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τρίτες χώρες για να δουν δηλαδή και να κατανοήσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ώστε να υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της ποσόστοσης. Και νομίζουμε ότι αφού ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις, τότε θα είμαστε σε θέση κατά πάσα θενότητα πριν της Παναγιάς του χρόνου να τροποποιήσουμε την τρέχουσα διαχείριση αυτών των πολύ συγκεκριμένων ποσοστώσεων. Αυτά θα μπορούσα εγώ να πω προς το παρόν σύντομα και είμαι και έτοιμος να δεχτώ ερωτήσεις αν έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ Περνάμε στη συζήτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις για την εκτελεστική αυτή πράξη για τη διαχείριση των δεσμολογικών ποσοστώσεων. Ο κύριος Φλάναγκαν ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Φλάναγκαν. Thank you Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω μεγαλύτερη ανησυχία στη χώρα μου όσον αφορά το θέμα αυτό για τις 78 τόνους μοσχαρίσιου ε, κράτος το οποίο είναι ημικατεψυγμένο και ημιφρέσκο έχει να κάνει με τις ψηλές τιμές τα τεμάχια. Τα για να καθιερώσουμε αν αυτό θα ισχύει. Ο καλύτερος τρόπος να το μάθουμε είναι να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις αγορές. Και συζητώντας εδώ ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν 150.000 τόνοι ήδη που εισάγονται Θέλουμε να δούμε τι είδη τεμαχίων έρχονται, γιατί ήταν ένας καλός δείκτης ε, για να μπορούμε να τα φιλτράρουμε όλα αυτά. Μπορείτε να μας ε, απαντήσετε σε αυτό, γιατί δυσκολεύομαστε να βρούμε τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο. Α, ο κύριο Μπούντα, συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Μπούντα.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 το θέμα δεν είναι να μιλήσουμε μόνο για τις ποσότητες ε, ή τις δεσμολογικές ποσοστώσεις ή ε, το ύψος των ε, εισαγόμενων προϊόντων, το, τις ποσότητες δηλαδή, αλλά να μιλήσουμε για την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλές όρους και προϋποθέσεις και υψηλές προδιαγραφές που επιβάλλουμε στους γεωργούς μας ως προς την εκλασιμότητα του κρέατος, ως προς τη χρήση των αντιβιωτικών ενώ ταυτόχρονα εισάγουμε προϊόντα που προέρχονται από δικαιοδοσίες με πολύ πιο χαλαρή νομοθεσία και παρόλα αυτά συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες με τέτοιες χώρες ή περιφέρειες. Θα πρέπει να εισάγουμε προϊόντα που πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές, τα ίδια πρότυπα και τους όρους που επιβάλλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους δικούς μας γεωργούς και κτηνοτρόφους. Γιατί πρόσφατα είχαμε το σκάνδαλο με βόλιο κρέας από τη Βραζιλία που έφτανε αλλοιωμένο, σάπιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει όχι μόνο η ποσότητα των εισαγωγών, αλλά και η ποιότητα, ιδιαίτερα στο κρέα. Ευχαριστώ κύριε Νόιχλου. Μια σύντομη ερώτηση. Αν είναι λογικό να γίνεται αυτή η εισαγωγή και η ερώτηση ότι όλοι μας ξέρουμε ότι το εμπόριο θα πρέπει στο μέλλον να είναι διαφορετικό, να διαμορφωθεί διαφορετικά και να μην σημαίνει ότι θα εισάγουμε μόνο τρόφιμα. Άρα η Επιτροπή έχει αναλογιστεί ποιος είναι ο σκοπός αυτού του είδους ε, εμπορίου. Ευχαριστώ. Αγγουλέρα. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί μου δημιούργησε κάποιες αμφιβολίες με την παρουσίαση που μας έκανε. Μας είπε ότι έχουμε 35 κανονισμούς ισχύ που καλύπτουν ε, όλο το κανονιστικό πλαίσιο για το θέμα αυτό. Και μάλιστα πρόκειται να τροποποιηθεί αυτό το σύστημα, γιατί δεν ε, εφαρμόζεται παρόμοια σε όλα τα κράτη-μέλη το κανονιστικό αυτό πλαίσιο και μας είπε ότι στόχος μας είναι η ενοποίηση και η εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου. Τι εννοείται, ότι παρόλο που υπάρχουν κανονισμοί που προβλέπουν τη διαχείριση του συστήματος αυτού με βάση το τελωνίο εισαγωγή, ε, ανάλογα με το τελωνίο εισαγωγή, η εφαρμογή είναι διαφορετική ε, και γι' αυτό χρειάζεται εναρμόνιση, γιατί αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, θα εισαγωγή θα προτιμούσα συγκεκριμένα πιο ευνοϊκά τελωνία εισόδου αν υπάρχει διαφοροποιημένη εφαρμογή. εκτό αν δεν κατάλαβα καλά την παρέμβαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν κρίνετε σκόπι με την εναρμόνιση σημαίνει ότι έχετε διαπιστώσει άνηση εφαρμογή, διαφορετική εφαρμογή. Ε, η... Ανάλογα με το τελωνίο ή τη χώρα εισόδου η διαχείριση είναι διαφορετική και άρα οι δασμοί που επιβάλλονται είναι διαφορετικοί. Θα ήθελα να μας το διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, δεν ζητά άλλο κανεί το λόγο από την Ομίγυρη, οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα που τέθηκε για την πρόσβαση στις πληροφορίες, και τη χρήση αυτών των ε, ποσοστώσεων, των δοσμολογικών ποσοστώσεων. Έχουν ήδη δημοσιευθεί αυτές οι πληροφορίες και μπορείτε να τις βρείτε όλες στην ιστοσελίδα της Ταξούντ, ε, της ε, DG Agri. Οι οικονομικοί παράγοντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα επικαιροποιημένο ε, σύστημα και γι' αυτό το λόγο στην DG Agri εργαζόμαστε σε ένα σύστημα πιο φιλικό προς το χρήστη, αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσια προσβάσιμες. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε για την εφαρμογή των γεωμικών προτύπων είναι ξεκάθαρο ότι οι τελωνικές αρχές των κρατών μελών ελέγχουν όλα αυτά τα γερμικά πρότυπα και τα πρότυπα αγοράς είναι καθήκον των κρατών μελών και μπορώ να σε διασφαλίσω ότι εφαρμόζονται ορθά. όσον αφορά αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε αυτόν τον καιρό και συγκεκριμένα τη διαδικασία εναρμόνισης. Μερικές από αυτές τις ποσοστώσεις ε, διαχει, τις διαχειριζόμαστε σε εβδομαδιαία βάση, μηνιαία βάση ή τριμηνιαία βάση σε συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα απλοποιήσουμε το σύστημα και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε κάποιες ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν καλοί λόγοι να ε, προχωρήσουμε σε μηνιαία διαχείριση. Ένα άλλο παράδειγμα, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε τα, τις ε, για άδεια εισαγωγής δεχόμαστε ότι κάποιος είναι οικονομικός παράγοντας παρέχοντας ένα, μια απόδειξη μπορεί, ένα proof of trade. Δηλαδή, ένα επίσημο έγγραφο που να δείχνει ότι τα προηγούμενα δύο έτη έχεις εισαγάγει τουλάχιστον 25 τόνους κάποιου προϊόντος. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, το ποσό μπορεί να είναι 50 τόνοι, 250 τόνοι. Έτσι μετά από συζητήσεις με την εφερόμενα μέρη συμφωνήσαμε για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία θα εφαρμόσουμε το ποσό των 25 τόνων. Ένα παράδειγμα απλοποίησης και εναρμόνισης που προσπαθούμε να πετύχουμε και μόνο όταν υπάρχουν καλοί λόγοι θα τηρήσουμε κάποιες τομεκές διατάξεις όπως είναι στην περίπτωση γαλακτοκομικών ποσοστώσεων όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Η κυρία Νόιχελ διαμαρτύρεται ότι δεν έλαβε απάντηση. Δυστυχώς η δική μου ερώτηση δεν απαντήθηκε. Παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτησή σας. Αν είναι νο... Ε, ε, λογικό να εισαγάγουμε από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη άκρη του κόσμου ε, κρέας όταν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση με τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να σκεφτούμε το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το εμπόριο μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρακαλώ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σύντομα. Σα ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ε, νόμιζα ότι κάνατε περισσότερο παρατήρηση, όχι ερώτηση ή δήλωση παρά ερώτηση. Είναι σαφές ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό. Οπότε και η λύση που θα πρέπει να βρεθεί σε αυτό θα πρέπει να είναι πολιτικής φύσης και όχι τεχνικής. Καλύτερα την ερώτησή σας να την παραπέμψετε στον συνομοθέτη, δηλαδή στην Επιτροπή σας, που συμμετέχει στη διαμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά. Ήταν κάπως γενική και όριστη απάντησή σας, αλλά δεν ήταν δυνατόν να δώσετε κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Οπότε, αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 5 και να καλωσορίσω θερμότατα τον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, τον κύριο Σάνι. Το αφήνω λίγο χρόνο να φορέσει τα ακουστικά του. Είχαμε τη συζήτηση των ε, τροπολογιών στις 16 του μηνός και μάλιστα είχαμε προβλέψει ότι στι 4 θα αρχίσουμε την ψηφοφορία, γι' αυτό καθυστέρησε κάπω ο εισηγητή. Κανονικά είπαμε η ψηφοφορία να ξεκινήσει στι 4, αλλά μια και στο μεταξύ ήρθε ο αρμόδιος εισηγητή, μπορούμε να ξεκινήσουμε και 5 λεπτά νωρίτερα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα τον κύριο Σάνι να μα κάνει την εισαγωγή για το θέμα αυτό του, της ετήσιας έκθεσης για την πολιτική του ανταγωνισμού. Μία σύντομη εισαγωγή παρακαλώ από τον εισηγητή μας τον κύριο Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω σύντομη για την έκθεση αυτή. Όπως ξέρετε, ε, το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του προβληματισμού μας στο θέμα της πολιτικής ανταγωνισμού και αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στον τομέα της γεωργίας και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει και αναγνωρίζει πια ότι η γεωργία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη ε, οποιοδήποτε άλλος κλάδος της ε, οικονομίας γιατί έχει ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία χρόνια είχαμε καταλήξει στην κατανόηση και την αντίληψη ότι η γεωργία και η γεωργική παραγωγή δεν χρησιμοποιούν κατάλληλα όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και από κοινού με τους και προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτές τις δυνατότητες για να τις αξιοποιήσουν καλύτερα οι Γεωργοί. Καταλήξαμε σε τελικά σε 16 συμβαστικές τροπολογίες και συμφωνήσαμε σε αυτές όλοι οι σκιώδεις ηγετές. Τους ευχαριστώ θερμά λοιπόν για την συνεργασία και ευελπιστώ ότι θα εγκριθεί η έκθεση και η συνεννόηση στην οποία κατέληξαν οι σκιώδεις θα αντικατοπτριστεί και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Πολύ σημαντική η ενημέρωση που μας κάνατε ότι υπήρχε συμφωνία για όλες τις συμβαστικές τροπολογίες με τους σκιώδεις ηγητές. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία θα ήθελα να σας πω ότι τα θέματα της διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων ε, τα συζητήσαμε με πρωτοβουλία της κυρίας Ράιρ, της συντονίστριας. Οι συντονιστέ ενέκριναν το αίτημά τη να ζητήσουμε εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, κάτι που έγινε στην προηγούμενη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάντω την κυρία Σράιερ, Πύριξ Ράιερ, για την πρωτοβουλία τη. Και περνάμε στην ψηφοφορία του σημείου 5 που προβλέπει την ετήσια έκθεση της πολιτικής ανταγωνισμού ακούσαμε μια σύντομη εισαγωγή από τον ε, εισηγητή μας και μια και ήρθε η ώρα 4 η ώρα της προγραμματισμένης ψηφοφορίας μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν ήθελα να ξεκινήσουμε νωρίτερα την ψηφοφορία για να προλάβουν να έρθουν όλοι οι ευρωβουλευτές για να ψηφίσουν. Παρακαλώ, ετοιμάστε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, γιατί τις ε, συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 9. Ε, ναι, περιμένουμε τον κύριο Ταραμπέλα να ψηφίσει. Οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 9. Ε, ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισε και ο κύριος Ταραμπέλα, άρα μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο κατά. Ελπίζω ρεμίτα του κύριου Ταραμπέλα. Πάμε στην τροπολογία 38 της κυρίας Δελαέ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μου λίγο αφηρημένος και δεν κατάλαβα το αποτέλεσμα. Στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 38 να με συμπαθάτε για την αφηρημάδα μου. Τέλος ψηφοφορίας. Μάλλον ε, είναι υπέρ ε, οι συνάδελφοι. Ναι, όντως. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά εγκρίνεται 77 υπέρ εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 6 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία τέλος Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική 13, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ εγκρίνεται. 16 υπέρ, εγκρίνεται. 17 υπέρ, εγκρίνεται. 18 Ποιος είναι υπέρ Κατά Εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε Καλύτερα έρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. με μία ψηφοδιαφορά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Άρχιτη ψηφοφορία, συγγνώμη, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται και πάμε στην ψηφοφορία του συνόλου της γνωμοδότησης μετά την, μετά την αποδοχή των τροπολογιών ηλεκτρονικά και η τελική ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κύριου Σάνη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε θερμά τον εισηγητή μας, τους και εισηγητέ και τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην διεκπαιρέωση αυτή τη γνωμοδότηση. Κύριε Σάνη, θέλετε το λόγο για οτιδήποτε. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Οπότε στις 4.30 έχουμε την ακρόαση, την κοινή ακρόαση των τριών επιτροπών, Άγκρι, Έμβη και Ήτρε, για την δασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως ε, ένα 20 μέχρι τις 4.30, οπότε Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά σας θέλουμε παρακαλώ στις 4.30 να επιστρέψετε στην αίθουσα.